όλων των, συναδέλφων και άρα θα είναι και περισσότερο αποδεκτή από όλους στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μάντερς. Τελειώνει άρα η συζήτηση. Η ίσοφορία θα γίνει αύριο στις 12.30 ώρα. Επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ε, προφορικές ερωτήσεις ε, στην Επιτροπή που αφορούν τα τεστ κοπόσεως των Ευρωπαϊκών Τραπεζών. Και να δώσω τον λόγο στην κυρία Βόρτμαν Κόλ Πορταπόλα ως μίας εθνοσυντακτών. could you please speak with the microphone? Το μικρόφωνο παρακαλώ. With the microphone. It's in the microphone. The microphone is working. Okay. Dit heeft commissaris Barnier. να καθίσει και ο κύριος Μπαργκέ. Κύριε Πρόεδρε, το ΕΛΚ ανησυχεί για τα ευρωπαϊκά τεστ αντοχής για τις τράπεζες που θα λάβουν χώρα τον Ιούνιο. Γιατί πέρσι ήταν αναξιόπιστα τα τεστ. Και το αποτέλεσμα το είδαμε στις Ιρλανδικές τράπεζες που πέρασαν τα τεστ μια χαρά και μετά βρέθηκαν σε σοβαρά προβλήματα. Αυτό πρέπει λοιπόν να αλλάξει. Το ερώτημα είναι το εάν ο δικός μας, ο τραπεζικός τομέας μπορεί να αντιμετωπίσει τα δύσκολα. Και έτσι θα πρέπει άρα να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στον τομέα αυτών. Εξού και το ερώτημά μου εδώ πέρα. Ποιες είναι οι σημαντικότερες αλλαγές που θα φροντίσουν να μην έχουμε την περσινή αποτυχία των τεστ αντοχής. Κύριε Πρόεδρε, πέρσι κάθε χώρα αποφάσιζε μόνη της ποιες τράπεζες θα υποστούν τα τεστ αντοχής. Αλλά τώρα η νεοσυσταθήσα Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή αποφάσισε πως τα κριτήρια θα είναι ίδια για όλες τις τράπεζες σε όλες τις χώρες. Και βεβαίως θα το τεστ αυτό θα είναι και τεστ και για τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές. Και ξέρετε σε κάποιες χώρες ε, ε, είχαμε μια επιτυχία του ποσοστού 85% σε άλλες χώρες ένα 50% του τραπεζικού τομέα. Δεν είναι επαρκές αυτό, οπότε θα ήθελα να μου το εξηγήσετε κύριε Πρόεδρε. Για τράπεζες διασυνοριακές χρειαζόμαστε έναν εύρωστο ευρωπαϊκό μηχανισμό ε, επίλυσης κρίσεων και άρα Μπορεί να έχουμε και άλλες τράπεζε σε κρίση, αλλά δεν επιτρέπεται πλέον να μην έχουμε μηχανισμό αντιμετώπισης της. Οπότε το ΕΛΚ θέλει να καταθέσετε φιλόδοξε προτάσεις και θα έχετε τη στήριξή μα εντό του Κοινοβουλίου. Σα ευχαριστώ. Κυρία Βόρτμαν Κόλ. Μια άλλη επίση συντάκτη για τρία λεπτά, η κυρία Μπόουλ. Κύριε Επίτροπε, η επίλυση τη τραπεζική κρίση ε, γίνεται σε διεθνέ επίπεδο και υπάρχουν και πολύ σημαντικά ζητήματα ανταγωνισμού που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αυτό δεν σημαίνει όμω ότι θα πρέπει όλα να περιμένουν, ειδικότερα όταν έχουμε και τραπεζική χρήση και ε, κρίση δημόσιου χρέους. Ε, το είχαμε ξαναπεί και την προηγούμενη εβδομάδα και το επαναλαμβάνουμε ότι οι δοκιμές αντοχής των τραπεζών θα πρέπει να είναι και σταθερές και διαφανείς και ε, αξιόπιστες. Θα πρότεινα λοιπόν να διδαχθούμε από τη ΣΥΠΑ και τον Ντόρτ Φρανκ που ζητάει ε, δημοσιοποίηση για δύο χρόνια και μιλάει για τις προβλέψεις ρευστότητας. Υπάρχουν ευρωπαϊκά ονόματα μέσα σε αυτές τις ε, αποκαλύψεις και καλό θα ήταν να κάνουν το ίδιο και οι ευρωπαϊκές ε, τράπεζες να προβούν σε αντάλογες αποκαλύψεις για το 2008-2009. Σε σαν συμπλήρωμα αυτών των stress test. Τώρα αυτές οι νέες δοκιμές έχουν βελτιωθεί ε, υπό την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών αλλά υπάρχουν και κάποιες ε, κολυσιεργίες από τα κράτη-μέλη και θα πρέπει να περάσει πια το μήνυμα ότι αν δεν υπάρχει πολιτική βούληση δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στην κρίση. Και είναι πολύ πιο δαπανηρές και οι λύσεις. Γιατί να προσπαθήσουμε να κρύψουμε το πλήρες επίπεδο έκθεση τραπεζών σε χρέος όταν γνωρίζουμε ποια είναι η πραγματικότητα, οι περισσότεροι από εμάς και δεν αποτελεί δικαιολογία ε, να μην ε, ε, προχωρήσουμε με αυτές τις δοκιμές αν δεν είχαν χάσει την αξία τους, πολλά από τα προϊόντα θα είχαν απομακρυνθεί από τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών και δεν θα είχαν παραμείνει εκεί μέχρι να λήξουν. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε πληροφορίες, πρέπει να εκτιμήσουμε το τι γίνεται και στα βιβλία των τραπεζών. Αλλά υπάρχουν κάποιες ζωφερές ερμηνείες που ε, περιλαμβάνουν και κάποια κράτη-μέλη που μπορεί να πληγούν. Πολλές φορές ένοχες είναι οι αποπτικές αρχές και όχι και τα κράτη-μέλη. Ε, όταν ε, μάλιστα δεν προσπαθούν ε, να κρύψουν για να συγκαλύψουν κάποια πράγματα. Κάποια κράτη-μέλη βέβαια λαμβάνουν μέτρα, πιέζουν τις τράπεζες να συλλέξουν περισσότερους σπόρους. Αλλά την υποκεφαλαιοποίηση δεν έχει σκεφτεί κανείς πώς θα την αντιμετωπίζει. Αν διδαχθήκαμε κάτι από την κρίση είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διασύνδεση και αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των τραπεζών και αν παγώσει η διατραπεζικός δανεισμός θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να υπάρχει συντονισμός ε, και αποκάλυψη των απαντήσεων. Αλλά δεν μπορούμε να χωρέσουμε έναν ελέφαντα μέσα σε ένα δωμάτιο, διότι δεν μιλάμε μόνο για τις τράπεζες, ε, μιλάμε για το δημόσιο χρέος, μιλάμε για τη σταθερότητα του ευρώ, τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους και πάρα πολύ σημαντικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα ο τελευταίος ε, συντάκτης ερώτησης, ο κύριος Σάντης Πρεσέδο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, είναι ώρα να έχουμε διαφανείς δοκιμασίες αντοχής που θα είναι και ευέλικτες και αξιόπιστες και αποτελεσματικές η ποιότητα, η εξοπιστία είναι σημαντική γιατί θα συμβάλλει στη χρηματοοικονομική σταθερότητα και στην εμπιστοσύνη των αγορών. Αυτές οι δοκιμές είναι ένα πολύ σημαντικό εποπτικό εργαλείο για την αξιολόγηση της φερεγγιότητας των μεμονωμένων τραπεζών, την αντοχή, την ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος συνολικά με το σχεδιασμό τους, με την άσκησή τους ε, θα δούμε πώς θα τα πήγαιναν οι τράπεζες ε, υπό ακραίες καταστάσεις και αν θα μπορούσε να αποφευχθεί ένα αποτέλεσμα ντόμινο, μια επιμόλυνση που θα οδηγούσε σε κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος. Έχουν γίνει από την Επιτροπή ε, των Ευρωπαίων Εποπτών κάποιες δοκιμές, η πρώτη το Μάιο του 2009, οπότε και το ΕΚΟΦΗΝ ζήτησε από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών τραπεζικής εποπτείας να εποπτεύσει αυτά τα stress test του χρηματοπιστωτικού συστήματος για να υπάρχουν συνολικά στοιχεία και πληροφορίες για την ανθεκτικότητα του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος συνολικά. Και επικεντρώθηκε στους 22 μεγαλύτερους τραπεζικούς ομίλους, αλλά δεν έγιναν γνωστά στο ευρύτερο κοινό τα στοιχεία αυτών των δοκιμών αντοχών. Απλά μια μεθοδολογία ε, αποκαλύφθηκε για τρία σενάρια, το καλύτερο, το ε, λιγότερο άσχημο και το χειρότερο, αλλά τελικά δεν υπήρξε πλήρης διαφάνεια. Τώρα, υπήρξαν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε τον Ιούλιο του 2009 η Κομισιόν για τις κρατικές ενισχύσεις, που έλεγε ότι οι τράπεζες που ε, έχουν ανάγκη από βοήθεια για να αντιμετωπίσουν την κρίση θα έπρεπε να υποβληθούν σε stress test. Την 1η Οκτωβρίου του 2009 τα συνολικά αποτελέσματα δόθηκαν, έγιναν γνωστά στο ΕΚΟΦΗΝ και στις 2 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους η ΣΕΠΣ, η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Υποπτίας ε, ζητήθηκε να εκπονήσει και νέα στρεστές μεταξύ άλλων, τα οποία ε, τα έκανε αυτή η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Υποπτίας και είχαν κάποια αποτελέσματα τα οποία δημοσιοποιήθηκαν ε, μετά από τις κατευθύνσεις ε, του Συμβουλίου του Ιουνίου 2010 και αφορούσαν 91 τράπεζες ε, στην Ευρώπη. Ασκήθηκε κριτική για το ότι ε, υπήρξε ευρωπαϊκή εστίαση, αλλά και γιατί κάθε χώρα αποφάσισε ποιε τράπεζε θα υποβληθούν ε, στι δοκιμέ αυτέ, γιατί είναι διαφορετική κατάσταση σε κάθε χώρα και δεν είχαν δοθεί και οι ε, ορθέ πληροφορίε πάντα, όπω παραδείγματο χάρη έγινε με την Ιρλανδία. Ή κάποιε τράπεζε σε κάποιε χώρε δεν έδωσαν τα πλήρη στοιχεία για το δημόσιο χρέο. Οπότε δεν μπόρεσε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπό τι συνθήκε αυτέ έχει φτάσει λοιπόν τώρα η στιγμή να έχουμε ένα νέο γύρο τέτοιων δοκιμών αντοχή. Αλλά είναι τελείω διαφορετικά τα πράγματα εδώ. Έχουμε νέε εποπτικέ αρχέ ευρωπαϊκέ. Για πρώτη φορά έχουμε αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο εποπτεία ε, βλέποντας τις δύο προηγούμενες πρακτικές και έχοντας αντλήσει τις εμπειρίες πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια τώρα, μεγαλύτερη αξιοπιστία και βέβαια μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα που είναι και το ουσιώδες στην τρίτη αυτή, στον τρίτο αυτό γύρο δοκιμών αντοχή. Θέλουμε να δούμε λοιπόν πώς θα αποφευθούν ε, τα λάθη των δύο προηγούμενων γύρων. Πρώτον και δεύτερον ε, τι θα γίνει για να γίνει αντιληπτός ο κίνδυνος που υπάρχει στα κράτη-μέλη, να γίνει δηλαδή κατάλληλη διάγνωση των κινδύνων. Κύριε Επίτροπε, επίσης πρέπει να δούμε ποια μέθοδος θα αναπτυχθεί σύμφωνα με τις διάφορες ε, μεθόδους διαπραγμάτευσης και τις τραπεζικές δομές. Άρα αυτές οι δοκιμές αντοχής θα πρέπει να μπορούν να δώσουν ε, τις αναγκαίες πληροφορίες για να υπάρξει και η ανάλογη αντίδραση. Θα πρέπει να δούμε και με τις νέες εποπτικές ε, αρχές τι θα γίνει. Παραδείγματο χάρη, στις 18 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών δημοσίευσε ένα πολυσέλιδο έγγραφο για τη μεθοδολογία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου, θέλω να δω, Κόπτεται ο ε, ε, Σας ευχαριστώ κύριε Σάντσες Πρεσέδο. Ακολουθεί ο Επίτροπος ο κ. Μπανιέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Κορίνα Βόρταν τον, και τους άλλους, τον Ζαν Πολ και τη Sharon Bowles για, την, ε, για την, τις ερωτήσεις τους που αφορούν την αξιοπιστία ε, των ε, δοκιμών αντοχής των τραπεζών. Θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Κύριε Πρόεδρε, η χρηματοπιστική βιομηχανία ανορθώνεται σιγά σιγά, έστω και για κάποιες τράπεζες θεωρούμε ότι η κρίση έχει τελειώσει. Τέλος πάντων, η κρίση αυτή ήταν δίαιη θα έλεγα ε, εμείς προσπαθούμε να εξάγουμε στα συμπεράσματά μας. Και αυτό χρειάζεται προσπάθεια. Για να συνειδητοποιήσουμε την κρίση και τα διδάγματα χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο επίβλεψης που το έχουμε από την 1η Ιανουαρίου χάρη σε εσά κυρίως. Χρειαζόμαστε εργαλεία πρόβλεψης, μια καλύτερη διακυβέρνηση σε κάθε ένα ίδρυμα. Χρειαζόμαστε επίσης μια καλύτερη κεφαλιοποίηση, θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό, και επίσης χρειάζεται να μετρήσουμε, να ε, σφιγμομετρήσουμε, να δούμε την θερμοκρασία ε, ανα πάσα στιγμή της βιομηχανίας αυτής. Γι' αυτό χρειαζόμαστε εργαλεία αξιόπιστα και οι δοκιμές αντοχής είναι ένα εργαλείο κλειδί σε αυτόν τον τομέα και το συζητήσαμε όχι μόνο εδώ αλλά και τον Απρίλιο με τους Υπουργούς Οικονομικών στα πλαίσια του Συμβουλίου. Όπως υπενθυμίσατε, πέρυσι οι δοκιμές αντοχής ήταν ανεπαρκείς, σαφέστατα. Και η Κομισιόν το είπε πάρα πολλές φορές και το είπε στη νέα αρχή επίβλεψης, στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, που συντονίζει τα, τις δοκιμές, τα τεστ σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές. Γι' αυτό θα πρέπει να διορτηθούμε για την ποιότητα και κυρίως για την αξιοπιστία των νέων δοκιμών του 2011 που ξεκίνησαν πριν μερικέ ομάδες τον Απρίλιο και θα απαντήσω στην ερώτησή σας και θα σας πω ποια είναι η ανάλυση μας και αυτό σε πέντε σημεία. Καταρχάς οι δοκιμές ε, για το 2011, όπως το επιθυμήσατε, βελτιώθηκαν σημαντικά και ουσιαστικά, κυρίως σε έξι σημεία που θα σας αναφέρω τηλεγραφικά. Το ένα αφορά το μακροοικονομικό σενάριο, το αντίθετο αν θέλετε, το οποίο προσωμιώνει ε, συνθήκες πολύ πιο δύσκολες από ό,τι το 2010 και αναφέρεται επίσης ε, και σε κρίση στον χρηματοσυμμετικό τομέα αλλά επίσης και τις συνέπειες στο κόστος χρηματοδότησης. Δεύτερον, η συνοχή ε, της όλης άσκησης ενισχύθηκε και στην αρχή αλλά και υπάρχει και μία ε, πιστοποίηση εκ των υστέρων. Τρίτον, ε, εφαρμόσαμε μία αρχή διαφάνειας, μία διευρυμένη αρχή διαφάνειας και τα αποτελέσματα του Ιουνίου θα ενισχυθούν αυτό και θα ε, συνοδευθούν με έναν απολογισμό των τραπεζών, κυρίως όσον αφορά το δημόσιο χρέος και την δομή του κεφαλαίου. 4. οι τράπεζες δοκιμάζονται με βάση ενώ ένα κατόφλι ανώτερου, ανώτερο ε, κατόφλι κεφαλαίου. 5. Ε, η διαμοσίευση ε, των αποτελεσμάτων από, εξ αρχής βελτιώνει την, την όλη δοκιμασία και εν η συνεργασία των κυβερνητικών αρχών για την εφαρμογή λύσεων για τις τράπεζες που δεν θα σεβαστούν, ε, που δεν θα περάσουν τα τεστ αυτά όλα αυτά βελτιώνουν και ε, το όλο σύστημα και νομίζω ότι αποτελούν μια πρόοδο και βλέπουμε ότι μέσα σε μια χρονιά βελτιώνουμε πάρα πολλά ε, θέματα. Δεύτερη ε, διαπίστωση χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη σαφήνεια όσον αφορά το δημόσιο χρέος και μου θέσατε μια ερώτηση για την μεθοδολογία που εφαρμόζουμε στον τομέα αυτό, όπως είπε και η ερώτηση η κυρία Βόρτμαν Κόλ. Αυτή, αυτό το αντίθετο αν θέλετε σενάριο προβλέπει μια πάρα πολύ σημαντική δοκιμή όσον αφορά τις διακή τη διακύμαση του δημόσιου χρέους όσον αφορά και τη διακύμαση τη χρηματοδότησής του. Το σενάριο αυτό δεν περιορίζεται μόνο στη χρεοκοπία και στην αδυναμία ε, επιστροφής αποπληρωμής του δημοσίου χρέους. Ε, το διατηρούμε στο trading, trading book των τραπεζών το δημόσιο αυτό χρέος. Και υπάρχει μια επιλογή όμως η οποία έγινε φέτος. Ε, εδώ τα, ε, σας υπενθυμίζω ότι οι δοκιμές αυτές ναι μεν προσωμιώνουν ακραίες, αποτελούν προσωμείωση ακραίων καταστάσεων αλλά πιστευτών όμω καταστάσεων, όχι μια απίθανης κατάστασης. Γι' αυτό ε, πιστεύουμε, εύλογα πιστεύω, και αυτό το πιστεύουμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ότι είναι πολύ πιο ε, χρήσιμο σήμερα να μιλάμε για την έκθεση απέναντι στο δημόσιο χρέος έτσι όπως ε, αυτό εμφανίζεται στο χαρτοφυλάκιο των τραπεζών και στο χαρτοφυλάκιο των διαπραγματεύσεων. Με τον τρόπο αυτό η παρουσίαση θα είναι πολύ πιο λεπτομερής από ό,τι πέρυσι. Επίσης, τρίτη παρατήρηση. Μας επιστήσατε την προσοχή για την ανάγκη να εφαρμόσουμε με ένα πιο συνεκτικό τρόπο τα σενάρια των stress test σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ήταν, είναι πολύ σημαντικό και για την αξιοπιστία της, του ολοχηρήματος. Η Τραπεζική Αρχή καταβάλει σημαντικές προσπάθειες κάνοντας μια ε, πολύ αυστηρή πιστοποίηση των αποτελεσμάτων των τεστ και με τον τρόπο αυτό θα ε, εξασφαλίσουμε μια συνοχή στα ε, αποτελέσματα και θα υπάρχει και μια σύγκληση ε, για τον τρόπο με τον οποίο ε, τα αποτελέσματα των τεστ θα συμπεριληφθούν στην, σε μια μελλοντική αξιολόγηση. Υπάρχει και ένα άλλο ουσιαστικό στοιχείο που αφορά την συνοχή και αφορά την προσφυγή σε κοινούς, ε, σε κοινές, ε, σε κοινούς ορισμούς όσον αφορά το κατόφλι των, ε, της κεφαλαιοποίησης. Οι, οι πόροι, θα, όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Αρχή, θα εκτιμώνται με βάση τις διατάξεις της οδηγίας για το κεφάλαιο που λαμβάνει υπόψη ούτως ή άλλως και τα μοντέλο διαχείρισης το οποίο εφαρμόζεται στην Ευρώπη. Τέταρτη παρατήρηση μας ρωτήσατε για την διαφορά κάλυψης του τραπεζικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τραπεζική αρχή ε, ε, προσπάθησε να δημιουργήσει ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα και σε ε, εθνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο διατηρώντας όμως ταυτόχρονα και ένα, ένα τρόπο διαχείρισης και αντιπροσωπεύει η, τα stress test του 2011 ε, το 75% των ευρωπαϊκών τραπεζών όσον αφορά το ενεργητικό και το δείγμα δημιουργήθηκε έτσι ώστε να καλύπτουμε τουλάχιστον το 50% του συνολικού ενεργητικού των εθνικών τραπεζών. Και τώρα για την ερώτηση που έθεσε ο κύριος Σάντσες Προσέντο για τα διορθωτικά μέτρα, τα backstops τα οποία περιμένουμε από τις τράπεζες, μάλλον τα οποία ναι, περιμένουμε από τις τράπεζες που είναι σε δύσκολη θέση. Ε, οι τράπεζες αυτές θα πρέπει να υιοθετήσουν κάποια μέτρα έτσι ώστε να διορθώσουν τις αδυναμίες τους και θα πρέπει να απευθυνθούν στο ιδιωτικό τομέα και να υπάρχει μια άμεση χρηματοδότηση είτε από τις αγορές είτε πολλών στοιχεία του ενεργητικού τους. Και μόνο εάν Εάν τα μέτρα αυτά είναι ανεπαρκή, τότε θα δοθεί μια δημόσια ενίσχυση στις τράπεζες αυτές. Βέβαια, η δημόσια αυτή ενίσχυση πρέπει να συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά τις ε, κρατικές ενισχύσεις. Και ο συνάδελφός μου κ. Σαρμούνια ασχολείται με το θέμα αυτό. Και τα, οι τράπεζες που αποφελούνται από αυτές τις ε, βοήθειες θα πρέπει, και εφόσον θα πρέπει να υποβάλουν στην Κομισιό ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης ανάλογα με το πρόβλημά τους. Αρκεί βέβαια η παμικρατική ενίσχυση να σέβεται την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και που θα εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά της μακροπρόθεσμα. Επίσης ζητήσατε και μια πολιτική ανακεφαλαίωσης και αναδιάρθρωσης των προβληματικών ε, τραπεζών, όπω αναφέρεται και στην έκθεση Φερέιρα για την ε, διαχείριση των κρίσεων. Ξέρετε κύριοι βουλευτέ, ε, ότι μα απασχολεί θετικό πλαίσιο για την επίλυση των κρίσεων, για, τον, την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα και αυτό το οποίο θέλουμε είναι αυτοί οι οποίοι θα κάνουν την επίβλεψη να έχουν στην διάθεσή του κάποιε λύσει για αυτά τα διεθνή, για αυτά τα, για τους διεθνείς τα ιδρύματα, διεθνή ιδρύματα, να τους δώσουμε κάποια εργαλεία έτσι ώστε να μην δημιουργούνται κρίσεις και αυτές οι κρίσεις να μην μας οδηγούν σε καταστροφές. Δηλαδή θέλουμε να έχουμε μία πρόορη, ε, αν θέλετε, παρέμβαση, οι τράπεζες να πληρώνουν για τις τράπεζες και αυτές είναι προτάσεις τις οποίες θα υποβάλλω και στο Συμβούλιο των Υπουργών αλλά και σε εσά πριν από το τέλος του καλοκαιριού. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις, οι απαντήσεις που ήθελα να σας δώσω ε, σαν ε, στοιχεία στις τρεις απάντηση στις τρεις ερωτήσεις που ετέθησαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Ακολουθούν οι ομιλητές ξενόματος ομάδων. Γκοζές για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Όπω είπατε και εσεί ο ίδιο, οι περσινέ δοκιμέ αντοχή ε, δεν είχαν τα προεξοφλημένα αποτελέσματα και γι' αυτό θα πρέπει τα ίδια σφάλματα και τη ε, σχεδιασμού και τη υλοποίηση να τα αποφύγουμε. Θα πρέπει τα παιδιά έρευνε να είναι συνεπή και αντίστοιχα. Γιατί πώ θα γίνει εξυγίανση αν δεν έχουμε σωστή διάγνωση. Θα πρέπει οι κυβερνήσει να το έχουν επίγνωση, να το έχουν ε, συνειδητοποιήσει αυτό. Βέβαια, οι δοκιμέ αντοχή φυσικά και θα πρέπει να είναι ρεαλιστικέ. Τα στοιχεία τα οποία μα δώσατε που ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένα, νομίζω ότι μπορούν να μας καλύψουν και τώρα η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ασκώντας την εποπτεία και αναλύοντας τα αποτελέσματα των δοκιμών αντοχής, θα πρέπει να μας δώσει ένα πρώτο αποδεικτικό στοιχείο για το πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι. Θα πρέπει να οριστούν οι μελλοντικέ ανάγκε πιθανής ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών και να ληφθούν τα μέτρα τα οποία εσεί αναφέρατε. Αλλά θα πρέπει να διεξαχθούν αξιόπιστα αυτές οι δοκιμές αντοχές για να ηρεμήσουν οι χρηματοπιστωτικές αγορές και να πάψουν να επηρεάζουν οίκοι αξιολόγησης και να έχουν βέβαια όλα αυτά πολύ αρνητικές επιπτώσεις για όλη την οικονομία. Η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των δοκιμών αντοχής ίσως ε, να δώσει ένα τέρμα ή να μετριάσει την εξάρτησή μας από τους οίκους αξιολόγησης. Ε, οι εποπτικές αρχές δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να φροντίσουν να είναι επιτυχημένες οι δοκιμές αντοχής, να δώσουν αποδείξεις γι' αυτό. Και ολοκληρώνοντα την παρέμβασή μου, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σα, κύριε Επίτροπε, σε ένα πολύ σοβαρό, κατά την άποψή μου, γεγονό ότι η νομοθεσία που αφορά του οίκου αξιολόγηση που τέθηκε σε ισχύ δεν εφαρμόζεται. Οι αρχέ που έχουν καταθέσει αυτές τους φακέλους τους οι και αξιολόγηση δεν έχουν λάβει κανένα ε, σχετικό μέτρο. Έχουμε προβλέψει μια μεταβατική περίοδο με το να τεθεί, μέχρι να τεθεί σε ισχύ η ΕΣΜΑ, αλλά τελικά είναι σαν να μην έχει γίνει τίποτα μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γκοζές. Η κυρία Ποδηματά για δύο λεπτά κύριε πρόεδρε κύριε επίτροπε εάν σε κάτι γίναμε σοφότεροι στην ευρώπη με την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση είναι ότι η πλήρης διασφάλιση επαρκούς κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών μας ιδρυμάτων και η αποτελεσματική εποπτεία γύρω από το ύψος των κινδύνων που αναλαμβάνουν αποτελούν σημεία κλειδιά της συνολικής όχι μόνο χρηματοπιστωτικής αλλά και οικονομικής διακυβέρνησης η επάνωδος με έναν τρόπο μόνιμο και συνεκτικό της ευρωπαϊκής οικονομίας σε ρυθμούς ανάπτυξης περνάει υποχρεωτικά και μέσα από την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη λειτουργία του τραπεζικού τομέα και της γενικότερης αποκατάστασης της ομαλής λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος με όρους διαφάνειας αλλά και με όρους επιστροφής στο βασικό του ρόλο ως μοχλού χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας όπως αποδείχθηκε στην πράξη και όπως επεσήμαναν ε, διάφοροι ομιλητές τα περσινά τεστ αντοχής δεν πέτυχαν το στόχο τους να καταδείξουν δηλαδή ποιες τράπεζες έχουν την απαιτούμενη αξιοπιστία απέναντι στους καταναλωτές στους πιστωτές τους αλλά και στους εθνικούς ρυθμιστές στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. φέτος βρισκόμαστε σε μια διαφορετική κατάσταση τα τεστ αντοχής θα δρομολογηθούν από τη νέα εποπτική αρχή την ευρωπαϊκή αρχή τραπεζών και θα πρέπει με κάθε τρόπο να αποφύγουμε την περσινή αποτυχία και βασική προϋπόθεση γι' αυτό είναι η επιβολή κοινών κριτηρίων αξιολόγησης της αντοχής των τραπεζών ενιαία ως προς την ερμηνεία και την εφαρμογή τους αλλά και ευρεία ώστε να καλύπτουν τους διαφορετικούς κινδύνους της κάθε εθνικής αγοράς. κύριε επίτροπε αυτό αποτελεί ασφαλώς την πρώτη προτεραιότητα στη φάση των δοκιμασιών αντοχής. θέλω όμως να σημειώσω ότι σε ένα δεύτερο στάδιο μια πλήρως ουσιαστική προληπτική εποπτεία θα πρέπει να περιλαμβάνει και τους κατάλληλους εκείνους μηχανισμούς που θα αντιμετωπίσουν έναν ιδιαίτερα διαφανή μέχρι σήμερα τομέα αυτόν του σκιώδους τραπεζικού συστήματος. Σας ευχαριστώ για τρία λεπτά η κυρία Γκουλάρ. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας κύριε Επίτροπε. Πολλά υπόθηκαν για τη μεθοδολογία, απαντήσατε αναλυτικά εσείς. Αυτό που θέλω απλά να κάνω είναι μια σύντομη παρατήρηση για το τι θα γίνει μετά τις δοκιμασίες αντοχής ε, συμφωνώντας με αυτό που ο κύριος Γκοζές ότι δεν αρκεί να περνάνε κάποια νομοθετικά μέτρα, πρέπει να γίνονται και σεβαστά, να τηρούνται. Από τη δική μου πλευρά σε αυτές τις δοκιμασίες αντοχής βλέπω το συμπλήρωμα του πακέτου οικονομικής διακυβέρνησης. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε με το δημόσιο χρέος, αλλά αν δεν εξηγιάνουμε τον τραπεζικό τομέα δεν θα τα καταφέρουμε. Πολύ απλά θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε αυτό το οποίο θα γίνει, αυτά τα μέτρα backstop που λέμε σε άπτες στα ελληνικά και άπτες στις άλλες γλώσσες. Τι πρέπει να κάνουμε με τις τράπεζες Είχα παραστεί στην ακρόαση με Μέρβιν Κίνγκ και Άντρια. Ενρία, Ανδρέα Ενρία, αντιπροέδρους ε, ε, του, Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Ο Μέρβιν Κίνγκ συγκεκριμένα μας είπε πράγματα διασκεδαστικά. Θυμάστε και την περσινή διαπραγμάτευση, κύριε Επίτροπε, μας είπε ότι οι ρήτρε ε, διάσωσης ή διασφάλισης που θέλουν να προσθεθούν οι χώρες μέλη στο πακέτο της Κομισιόν, παρόλα αυτά δεν εμποδίζουν το να γίνουν σεβαστές οι ενδείξεις της Ευρωπαϊκής ε, Αρχής Τραπεζών σε ό,τι αφορά την επανακεφαλαιοποίηση. Αυτό το στοιχείο θέλω να το θέσω υπόψη σας. Από συστημικής πλευράς η, το ίδιο η Επιτροπή Συστημικού Κινδύνου θεωρεί ότι είναι σημαντικό και πιστεύω ότι αν η ποιότητα του έργου τη Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών με τη δική σα στήριξη, με τον έλεγχο τη Επιτροπή ε, Συστημικού Κινδύνου, επιτρέψει στο να εγκρίνουμε με τα χαρά αυτέ αυτές τις ρήτρε στο πακέτο εποπτείας θα έχουμε κάνει ένα βήμα προς τα εμπρό. Ελπίζω η Κομισιόν με την Επιτροπή στην Κινδύνου πραγματικά να φροντίσει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα από τα μεγάλα ή μικρά κράτη-μέλη. Ένα παράδειγμα μας δίνει η Ισπανία. μα δινει η ισπανια ελπιζω να ακολουθήσουν και άλλε χώρε. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Φόρντ επίσης για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Τα τεστ του περσινού καλοκαιριού υποτίθεται πως ε, θα ηρεμούσαν τις αγορές. Δεν επέτυχε αυτό. Μετά από εννέα εβδομάδες κατέρευσαν οι Ιρλανδικές τράπεζες και αναγκάστηκαν να τις διασώσουν οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι και μάθαμε πως 12 δισεκατομμύρια από την πορτογαλική διάσωση θα πάνε πάλι στι τράπεζε τους. Δεν έχει λυθεί αυτή η κρίση και δεν θα λυθεί μέχρι οι αγορές να δώσουν αρκετή ε, ρευστότητα στις τράπεζες. Οπότε τα τεστ αυτά θα πρέπει να τονίσουν τους κινδύνους για τους οποίους ανισχούν οι αγορές και αυτή τη στιγμή οι αγορές ανισχούν για το δημόσιο χρέος. Το να μην δοκιμάσουμε το δημόσιο χρέος σε όλους τους ισολογισμούς δεν θα αποκαταστήσει την ε, εμπιστοσύνη γιατί αυτή τη στιγμή η ευρωπαϊκή Ε, εποπτική αρχή βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση το να παραδεχτεί ότι υπάρχει κίνδυνος μείωσης αξίας αυτών των χρεογράφων ίσως ε, προκαλέσει ακριβώς τη μείωσή τους αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορεί και το να αρνείται και από την άλλη βεβαίως είναι το ζήτημα του είδους του κεφαλαίου που έχουν αυτές οι τράπεζες και όσο προχωράμε αντιλαμβανόμαστε όλοι πως δεν είναι όλες οι τράπεζες ίδιες και ανησυχούμε για ανησυχούν ε, οι αγορές. Αλλά πρέπει να δούμε βέβαιως και τον παρονομαστή αυτού του κλάσματος. Ποια είναι ακριβώς και τα στοιχεία ενεργητικού αυτών των τραπεζών και αν μπορούμε να τα εμπιστευτούμε. Καθώς εάν υπάρχει ανάληψη κινδύνου κατά 50% μεγαλύτερη στις αμερικανικές τράπεζες, μήπως επιτρέπουμε στι ευρωπαϊκές να μην παρουσιάζουν σωστά του ε, κινδύνου τους. Για τους δανειστέ λοιπόν και τους ε, φορολογούμενους δεν προσφέρουν τα τεστ αυτά διαφάνεια και αυτό αγαπητοί συνάδελφοι είναι παροδία. Ευχαριστώ κυρία Φόρτ Γκίγκολτ για 3,5 λεπτά. Ναι αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Μπαρνιέ, το θέμα αυτό των τεστ ε, των τραπεζών είναι αποφασιστικό και τον παρακολουθούν οι πολίτες γιατί οι τράπεζες είναι στο κέντρο αυτής της κρίσης. Επένδυσαν τα χρήματά τους χωρίς να δουν τον κίνδυνο και με έτσι σε κάποια κράτη-μέλη που τώρα βρίσκονται σε κρίση δημιούργησαν κρίση, φούσκες με ακινήτων και άρα έχουμε καταστάσεις τις οποίες ε, οι αγορές ε, γνωρίζουν και χειρότερα από πολλούς ε, άλλους παρατηρητές. Και με αυτόν τον τρόπο προκλήθηκε η κρίση. Και τώρα βλέπουμε πως επιπροσθέτως αυξήθηκε πάρα πολύ το δημόσιο χρέος. Πρώτα απ' όλα μέσω των τραπεζικών εγγυήσεων και βεβαίως μέσω της ύψης αυτής. Οπότε το ζήτημα είναι εάν θα βγάλουμε σοβαρά συμπεράσματα από αυτή την κρίση. Αλλά δεν είναι το ζήτημα μόνο της παρελθούσας ευθύνη των τραπεζών, αλλά και το ότι ακόμα δεν λειτουργούν σωστά οι ε, αγορές. Ξέρετε πως εντωμεταξύ έχουν συγκεντρωθεί άλλα 427 δισεκατομμύρια ευρώ σε ανοιχτές απαιτήσει μεταξύ των τραπεζών γιατί δεν λειτουργεί πλέον το διατραπεζικό σύστημα και έχουμε πάρα πολύ μεγάλες αδυναμίες άρα του τραπεζικού... Όχι, με συγχωρείτε. Λόγω ακριβώς αυτής της ε, αδυναμίας δεν τολμούμε να αναλάβουμε τα μέτρα εκείνα τα οποία χρειάζονται για την ελάφρυνση του χρέου Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιρλανδία. Και οι άνθρωποι εκεί πέρα υποφέρουν ακριβώ λόγω τη κατάσταση του τραπεζικού συστήματο. Και άρα τα προηγούμενα δύο χρόνια είχαμε τα τεστ αυτά και λέγαμε επιτέλου θα μάθουμε την αλήθεια. 2010 είπαν πολλοί συνάδελφοι, τα τεστ αυτά δεν ήταν αρκετά σκληρά, ειδικά όσον αφορά τα κρατικά ομόλογα, τα οποία δεν ελήφθησαν καν υπόψη ω ε, κίνδυνοι τώρα το 2011 κάτι ανάλογο και το είπατε κύριε Μπαρνιέ, είπατε αρκετά πράγματα, δεν μας είπατε όμως γιατί οι κίνδυνοι των κρατικών ομολόγων λαμβάνονται υπόψη στο trade book αλλά όχι στο bank book. Μιλάμε για φοβερή υπεκφυγή όσον αφορά την πολιτική ευθύνη εδώ πέρα. Αυτή η ε, ομπρέλα την οποία ανακοινώσατε δεν είναι κάτι το ε, αυτονόητο. Πρέπει να τον εγκρίνει το κοινοβούλιο γιατί εδώ πέρα έχουμε κοινωνικοποιήσει ιδιωτικούς κινδύνους που έχουν αναλάβει οι τράπεζες. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει επίσης και ανάλογο τρέστ και επιμένω εδώ πέρα για την αγορά των ασφαλιών και σας παρακαλώ να το κοιτάξετε κύριε Μπαρνιέ. Είμαι απογοητευμένος γιατί η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή η οποία είναι υπεύθυνη δημιουργήθηκε και δυστυχώς δεν πέρασε τα δικά της τα τεστ. Οπότε σας παρακαλώ κύριε Μπαρνιέ βλέπουμε το εξής από το, την ιστορία αυτή. Ο Μπέρτολτ Μπρέχτ είχε πει πως οι αγορές είναι πάρα πολύ χειρότερες από μια τραπεζική ληστεία. Είχε κάνει λάθος όμως. Το να αποκρύφτουμε τη χρεοκοπία είναι πάρα πολύ χειρότερο. Ευχαριστώ. Ο κ. Μέρφυ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Η ουσιαστική αδυναμία των προτινόμενων stress test θα αναφέρθηκε. Είναι η δυνατότητα να έχουμε... Ε, να έχουμε ε, διευρυμένες χρεοκοπίες το κράτος της Ιρλανδίας ε, χρωστάει 720 δισεκατομμύρια λίρες και ε, ανεξάρτητα από το κόστος και από, την, ε, και από το επιτόκια για, την, για τα δάνεια τα οποία μας δίνουν είναι σίγουρα ότι θα χρεοκοπήσουμε. ούτως ή άλλως όλες οι χώρες η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία ε, έχουν εκτεθεί και ε, ε, ούτως ή άλλως πολλές τράπεζες των υπολείπων κρατών της, της Ευρώπης είναι εκτεθειμένες σε ομόλογα των χωρών αυτών. Βέβαια αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να, σταθεροποιηθεί το τραπεζικό τομέα. Όμως 33 δισεκατομμύρια ευρώ ε, τα οφείλουν έξι ε, Ιρλανδικές τράπεζες και ε, Τίτε να χρηματοδοτηθούν, να ενισχυθούν από την Ευρωπαϊκή Αρχή, από, την το Ευρωπαϊκό Σύστημα ε, Ενίσχυσης των Τραπεζών. Ε, αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι ότι τα μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα δεν μπορούν να, περιμέ... παραμείνουν στα χέρια των ιδιωτών, διότι με τον τρόπο αυτό ε, οι πολίτες ε, ε, πληρώνουν ένα μεγάλο κόστος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θα πρέπει να τελειώσει η δικτατορία των ε, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Θα πρέπει ε, να δίνονται, να μπορούμε να, να δίνουμε δάνεια στους, ε, στους ανθρώπους, θα πρέπει να δίνονται στεγαστικά δάνεια κτλ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πάσκα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Δημοσιεύτηκαν πρόσφατα τα νέα σενάρια και η μεθοδολογία για τα stress test που θα ελέγξουν ε, την αντοχή των Ευρωπαϊκών Τραπεζών. Αν θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι τα αποτελέσματα θα γίνουν δεκτά και από του ειδικού, ε, δεν θα πρέπει να είμαστε επιφανειακοί αλλά ούτε και ασυνεπεί, όπω έγινε τον Ιούλιο του 2010 επειδή η αξιοπιστία ολόκληρου του χρηματοπιστωτικού τομέα της Ευρώπης ενδέχεται να κρυθεί από την ε, σοβαρότητα αυτών των δοκιμών αντοχή, θα πρέπει αυτές να είναι στο δυνατόν πιο πλήρης και να λάβουν υπόψη ε, του κινδύνου που ενδέχεται να αντιμετωπίσει σε τέτοιου καιρού σε τέτοιε εποχέ, ο χρηματοπιστωτικό τομέα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει και κατάλληλη αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο εκτίθεται, είναι εκτεθειμένες οι τράπεζε ε, στο δημόσιο χρέο ή στο χρέο άλλων τραπεζών, ώστε να δούμε τα πιο ε, δυσμενή, τα πιο αντίξωα σενάρια που μπορεί να υπάρξουν, όπω παραδείγματο χάρη η χρεοκοπία μια χώρα. Θα πρέπει να δούμε επίση ότι υπάρχουν διαφορετικέ επιχειρηματικέ πρακτικέ χρηματοπιστωτικές και τραπεζικές δομές ανάλογα με το κράτος μέλος. Θα πρέπει να καλύψουμε πλήρως τα κράτη-μέλη γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κερσία Μαργκάγιο δεν είναι εδώ, οπότε δίνω τον λόγο στην κυρία Φερέιρα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, στις δοκιμασίες αντοχής των τραπεζών το 2010 νομίζω ότι όλοι αναγνώρισαν ότι ένα από τα βασικότερα προβλήματα με τις τότε δοκιμασίες ήταν ότι εφαρμόστηκε εθνική λογική και σε ό,τι αφορά τη μεθοδολογία και σε ό,τι αφορά τη διάγνωση, την επιλογή των κριτηρίων δηλαδή. Στην έκθεση που είχα συγγράψει εγώ Ζητεί το Κοινοβούλιο ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης στη διαχείριση της τραπεζικής κρίσης. Όμως στο μεταξύ δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συστημικού Κινδύνου, συγκροτήθηκε και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Και τελικά όλα αυτά έδειχναν ότι πράγματι θα δινόταν στην τραπεζική εποπτεία μια ευρωπαϊκή διάσταση. Παρά τα αυτά, δοκιμασίες αντοχής τελικά περιγράφονται από το Συμβούλιο ότι θα πρέπει ε, να οδηγήσουν σε φιλόδοξες στρατηγικές με βάση τα αποτελέσματά τους ε, να δοθούν μάλιστα και λύσεις ιδιωτικού τομέα, αλλά να παρασχεθεί και ένα στέρεο πλαίσιο σύμφωνα με τους κρατικούς κανόνες για την κρατική υποστήριξη σε περίπτωση που αυτό καταστεί αναγκαίο. Τι κάνουμε δηλαδή τελικά αυτή τη στιγμή βλέπουμε να επανέρχονται οι δοκιμασίες αντοχής και πάλι μιλάμε για τα κράτη-μέλη και δεν υπάρχει κανένα εναρμονισμένο πλαίσιο. Φυσικά και πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εθνικές ιδιαιτερότητες, αλλά δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω στην εθνική διάσταση. Δεν πρέπει να αφήσουμε μόνο τα κράτη-μέλη να επιλύουν ε, και να διορθώνουν τα προβλήματα. Είναι θέμα αρχής αυτό το οποίο τίθεται με τέτοιου είδους μεθοδολογία χάνουμε μια χρυσή ευκαιρία. Γιατί θα μπορούσαμε να δώσουμε μια γνήσια ευρωπαϊκή διάσταση στην τραπεζική υποπτία. Δεν το κάνουμε όμως. Σε ευχαριστώ κυρία Φερέρα. Ο κύριος Σμιτ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ξέρετε πως η καιρή είναι δύσκολη, η οικονομική κρίση επηρεάζει τους πολίτες και αυτοί έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στις τράπεζες. Τα τεστ αντοχής λοιπόν των τραπεζών είναι σημαντικό μέσο για να αποδείξουμε την αντοχή των τραπεζών σε αναπάντεχα οικονομικά σοκ γιατί από εκεί εξαρτάται η οικονομική σταθερότητα. Οπότε αποτελεσματικά τεστ θα αυξήσουν την εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα. Αυτό το γνωρίζουμε εκ πείρας. Σκληρίες, αξιόπιστες δοκιμές με σαφείς απαιτήσει. Νομίζω πως το παράδειγμα της Ιρλανδίας εδώ πέρα αποδεικνύει ποιε είναι οι συνέπειες εάν δεν το κάνουμε αυτό. Θεωρώ λοιπόν πως θα πρέπει να δημοσιευτούν τα τεστ μεμονωμένα ανά τράπεζα και είναι σημαντικό αυτό για την εμπιστοσύνη των πολιτών. Όπως είπε και ο κύριος Μπαρνιέ, το θέμα είναι θέμα εμπιστοσύνης. Οπότε θα πρέπει να έχουμε σοβαρές απαντήσεις σε αυτά τα οποία επικρατούν στην αγορά και θα πρέπει να καλύψουμε και την έκθεση στο δημόσιο χρέος και νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, εάν είναι να βελτιωθεί η εμπιστοσύνη των αγορών η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συστημικού Κινδύνου θα πρέπει να φροντίσουν να υπάρξει συνέχεια αυτών των δοκιμών και να αξιολογήσουν σωστά τους κινδύνους. Κύριε Πρόεδρε, αν οι τράπεζες δεν μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτά τα κριτήρια και τις απαιτήσει, θα πρέπει να δράσουν τα κράτη-μέλη. Έχουμε δει τη σημασία των τραπεζών και έχουμε δει πόσο γρήγορα οι κίνδυνοι μεταβάλλονται σε πραγματικές ζημίες. Πρέπει να είμαστε λοιπόν πάρα πολύ προσεκτικοί. Μπορεί να είναι καταστροφικά τα αποτελέσματα εάν δεν λάβουμε τα παλέτα μέτρα. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά ο κύριος Λάμπερτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα γαλλικά. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, οι δοκιμασία αντοχής είναι το τελευταίο προϊόν ε, του σειρμού της μόδας. Έχουμε μια βαθιά οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Ωραία, θα υποβάλουμε σε δοκιμασίες αντοχής ε, τις ε, τράπεζες. Το ίδιο κάνουμε με τα πυρηνικά εργοστάσια λόγω της πυρηνικής κρίσης. Λες και Ακριβώς ο θεσμός αυτός, ε, η ίδια ιδέα περί ε, δοκιμασιών αντοχής ε, θα δώσει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη είτε στους πολίτες είτε στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Γιατί τα πάντα εξαρτώνται από τις υποθέσεις, από τα σενάρια. Και πράγματι τα περσινά stress test δεν μπορούμε να πούμε και τόσο αξιόπιστα κύριε. Επίτροπε και σε ό,τι αφορά και τα πυρηνικά stress test όπως είπε ο Επίτροπος Έτιγκερ το μεσημέρι είναι ένα αστείο μέχρι στιγμής διότι να υποθέσουμε ότι πέφτει ένα αεροπλάνο ε, πάνω σε ένα πυρηνικό σταθμό και εκρήγνεται είναι ένα σενάριο το οποίο καν δεν λαμβάνεται υπόψη. Ε, λοιπόν, πρέπει, λέμε, κύριε Επίτροπε, να λάβουμε ε, υπόψη μας κάποια σενάρια πιστευτά. Όχι ίσως δηλαδή τη χρονοκοπία ενός κράτους μέλους. Ε, τελικά, θεωρείτε ότι αυτό το σενάριο ε, δεν είναι δυνατό, γιατί αυτό σημαίνει ότι αρνείστε την πραγματικότητα. Αν δούμε τα στοιχεία για το ελληνικό χρέο ή το ιρλανδικό χρέο, είναι σαφέ ότι αργά ή γρήγορα είτε αναδιάρθρωση του χρέου θα κάνουν, είτε εσεί τελικά παίζετε με το χρόνο, παίζετε με το ρολόι. Γιατί όσο καθυστερήσει αυτό, τόσο πιο πολύ θα στοιχήσει, τόσο πολύ θα κοστίσει σε όλου μα. Θέλω λοιπόν να επιδείξετε ευθύνη και αίσθηση τη πραγματικότητα, ε, κύριε Επίτροπε, διότι είστε ένα ε, φιλόδοξο ε, Ευρωπαίο και αυτοί που τελικά ε, αποδεικνύουν την αντοχή τους καθημερινά είναι οι πολίτες μας και αν δεν πάρουμε τον ε, τάβρο από τα κέρατα δεν θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη είτε των χρηματοπιστωτικών αγών ούτε των συμπολιτών μας. Τι θα πει πιάνω τον ε, τάβρο από τα κέρατα, από τα κέρατα σήμερα. Κάνουμε την, όλη την αναδιάρθρωση που χρειάζεται αλλά πρέπει να έχουμε και ένα είδος δημοσιονομικής ομοσπονδοποίησης θα έλεγα. Αλλά αυτό μπορούμε να το ξαναδούμε μια άλλη φορά. Ευχαριστώ Κύριο Κάρας για δύο λεπτά. Κύριε Επίτροπε, κύριε μου και κύριοι, πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την αναλυτική απάντηση της κοινοβουλευτική μου ερώτησης για τα τεστ της ε, ερωτηση 8 Φεβρουαρίου. Διαπιστώνουμε εδώ πέρα όλοι πως το ζήτημα είναι η σοβαρότητα και η εμπιστοσύνη, η ειλικρίνεια και η αποφασιστικότητα και έτσι μπορούμε να ξεπεράσουμε την κρίση εμπιστοσύνης. Αλλά πρέπει να πω πως εγώ δεν τα βλέπω αυτά στα τελευταία stress tests. Η σωστή δηλαδή αξιολόγηση. Οι συνέπειες είναι άγνωστες, τα συμπεράσματα μας τα είπατε σήμερα και οι συνέπειες από τα επόμενα τεστ είναι ακόμα άγνωστες. Έχω λοιπόν τρία ερωτήματα. Πρώτον, πώς μπορείτε αυτή τη φορά να μας εγγυηθείτε κύριε Επίτροπε πως μιλάμε μακροπρόθεσμα και δεν εστιάζουμε μόνο βραχυπρόθεσμα όπως έγινε με τις Ιρλανδικές τράπεζες. Δεύτερον παρατηρούμε μπροστά στα μάτια μας επιδίνωση της κρίσης δημοσίου χρέους, τα είπε ο κύριος Γκίγκολτ, η επιδίνωση αυτή όμως θα εξεταστεί μόνο στα trade books των ε, τραπεζών και όχι στο bank book το οποίο δεν θα συμπεριληφθεί στα stress tests. Μήπως εδώ πέρα πάλι δίνουμε την αίσθηση πως υπάρχει η εγγύηση μακροπρόθεσμη ενώ δεν φωτίζουμε την πραγματική διάσταση του προβλήματος του δημοσίου χρέους. Ευχαριστώ κύριε Κάρας. Για δύο λεπτά ο κύριος Σάντσες Πρεσέδο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπο, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την απάντησή του. Το σημαντικό είναι να γίνει η σωστή διάγνωση και βέβαια μετά να γίνει και σωστή θεραπευτική αγωγή. Άρα μεγαλύτερη αξιοπιστία, μεγαλύτερη διαφάνεια των stress test, αλλά πρέπει να είναι αποτελεσματική και η ανταπόκριση. Πρέπει λοιπόν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί να είναι φερέγγοι, το χρηματοπιστωτικό σύστημα να είναι σταθερό και πάνω απ' όλα θα πρέπει να αποκαταστήσουμε και την, ε, την πιστωτική ροή ε, στην πραγματική οικονομία. Θα πρέπει να γίνουν όλες οι προσπάθειες για να αντιμετωπιστούν αντίξωα σενάρια από όλες τις τράπεζες και θα πρέπει να προετοιμαστούν οι τράπεζες όσες δεν περάσουν τις δοκιμασίες αντοχής να βρουν τα απαραίτητα μέτρα για να ξεπεράσουν το πρόβλημα και θα πρέπει τα κράτη-μέλη όσα δεν το έχουν κάνει ακόμη να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την επανακεφαλαίωση ή για να βρουν κάποια ζητήματα, να βρουν κάποιες λύσεις στο θέμα της εξυγένσεως των τραπεζών. Σε ό,τι αφορά τώρα την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών μπορεί να διατυπώνει συστάσεις, ε, μπορεί να εντοπίσει ε, πού υπάρχουν συστημικοί κίνδυνοι και μπορεί επίσης να παρακολουθεί και τις διαδικασίες ε, εξυγίανσης ή διάσωσης. Θα έχετε τη στήριξή μας, κύριε Επίτροπε, για να προτείνετε ένα φιλόδοξο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Θέλουμε περισσότερη χρηματοοικονομική ολοκλήρωση, κυρίως όμως φορολογική και πολιτική. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Σάντσες Πρεσέδο. Για δύο λεπτά ο κύριος Στόλογεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Τα τεστ αυτά είναι σημαντικά για να αξιολογήσουμε την υγεία του τραπεζικού συστήματος, αλλά πρέπει να εκπληρωθούν εδώ πέρα δύο κρίσιμες προϋποθέσεις να είναι επαρκώς ποιοτικά τα τεστ αντοχής και βεβαίως και η αξιολόγηση να είναι ακριβής. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω πως οι τράπεζες είχαν διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Στη Ρουμανία, όπως και αλλού, οι τράπεζες δεν είχαν μπλέξει με τοξικά λεγόμενα ομόλογα αλλά είχαν μια επέκταση της ε, ρευστότητα με βάση μακροπρόθεσμη ε, μακρο, με βραχυπρόθεσμους ε, πόρους. Το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο όμως, δηλαδή ζημίες και άρα βρέθηκαν σε πάρα πολύ ευάλωτη θέση και ε, δεν υπήρχε ανάληψη ευθύνης για την διαχείριση κινδύνου που έκαναν. Δεύτερον, χρειάζεται να είναι διαφανή τα αποτελέσματα των τεστ αυτών αντοχής. Οι αγορές και οι πολίτες το ζητούν, ζητούν διαφάνεια. Σας ευχαριστώ κύριε Στόλογιαν. Για δύο λεπτά ο κύριος Λούντβιξον. το τελευταίο έτος ε, αναταραχών στο χρηματοπιστωτικό τομέα νομίζω ότι χάσαμε ε, το επίκεντρο, τη ρίζα του προβλήματος. Προσπαθούμε να σώσουμε τις ε, πιο ευάλωτες χώρες και τα οικονομικά τους. Ξεχάσαμε όμως ότι το πρόβλημα ε, το έχουν οι τράπεζες. Από τη μια πλευρά έχουμε καταστροφές ε, με τα δάνεια στον τραπεζικό τομέα, εξού και τόσο τροτάται οικονομικά κάποιων χωρών, αλλά υπάρχουν ε, σημεία, αδύναμα σημεία στις τράπεζες, τα οποία εξακολουθούν να υφίστανται. Βλέπουμε οι λύσεις που προτείνονται στην Αθήνα, στη Λισαβόνα ή στο Δουβλίνο, ναι μεν υπάρχουν αλλά δεν φαίνεται να αποδίδουν αυτά αναμενόμενα. Εάν αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν καταβάλουμε την απαιτούμενη προσπάθεια για να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο, ένα αναϊφόρο τραπεζικό τομέα, αργά ή γρήγορα θα επιβαρυνθούν ε, τα κρατικά οικονομικά τόσο πολύ που δεν θα μπορούν ε, να επιβιώσουν τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη. Βλέπουμε ότι και οι χώρε που έχουν στιβαρά οικονομικά λίγα κάνουν για να αντιμετωπίσουν τι αδυναμίε του τραπεζικού του συστήματο. Φωνάζουν και ζητούν μέτρα από την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και την Ελλάδα, αλλά δεν κάνουν τα, ε, τη δική του ε, κατοίκον εργασία, θα έλεγα. Παρά τα προβλήματα τα οποία ε, είναι προφανή. Θα πρέπει σίγουρα να είναι σκληρές, διαφανείς και αξιόπιστες οι δοκιμές αντοχής, αλλά είναι προφανές ότι θα πρέπει να ακολουθήσει και η λήψη σοβαρών μέτρων για να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες που προανέφερα. Και θα ήταν πάρα πολύ πολύτιμη μια ευρωπαϊκή στρατηγική. Ελπίζω σύντομα να ε, προβεί στην σχετική πρωτοβουλία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί υπήρξε και η σχετική κατεύθυνση που δόθηκε από μια έκθεση του Κοινοβουλίου. Όλες οι χώρες, όχι μόνο οι ισχυρότερες, πρέπει να φροντίσουν, να επιλύσουν ε, και να κλείσουν ε, τις ε, μαύρες τρύπες που υπάρχουν στα τραπεζικά του συστήματα. Σας ευχαριστώ για ένα μισή λεπτό. Ο κύριος Μαν. Σας ευχαριστώ. Τα stress test των τραπεζών τα περσινά, ξέρετε κύριε Μπαρινιέ πως έπρεπε να είναι καλύτερα δεν φτάνει να μιλάμε μόνο για τα ίδια κεφάλαια, πρέπει να εξετάσουμε τις επιπτώσεις της κρίσης στη ρευστότητα των τραπεζών. Γιατί τότε κατέρευσαν τράπεζες όπως οι Lehman Brothers από προβλήματα ρευστότητας. Και δεν καταλαβαίνω τη συζήτηση για το εάν τα αποτελέσματα της εξέτασης ρευστότητας πρέπει να δημοσιοποιηθούν ή όχι. Όποιος θέλει να αποσιοποιήσει στοιχεία, τότε είναι σαφής η πρόθεσή του. Θέλει να εμποδίσει οι αγορές να μην σταματήσουν να εμπιστεύονται τις τράπεζες εκείνες που θα κοπούν στα τεστ. Όποιος θέλει λοιπόν να μην υπάρχει σαφήνεια για τα αποτελέσματα, τι κάνει. Θα οδηγηθούμε σε διασπορά φημών και μισών αληθιών. Θα πρέπει λοιπόν με τις μεθόδους και τις διάφορες παράμετρους, ο στόχος να είναι κοινό διαφάνεια για να δούμε πόσο αντέχουν στην κρίση οι ευρωπαϊκές τράπεζες. Χρειάζεται επιγόντως να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και προς το συμφέρον των ιδίων των τραπεζών. Ευχαριστούμε κύριε Μαν. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Κάντσιαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κάνετε μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Εμείς θα πρέπει να αποκτήσουμε, επανακτήσουμε σταθερότητα και εμπιστοσύνη. Για να γίνει κάτι τέτοιο, οι προσπάθειες πρέπει να είναι τεράστιες. Εσείς λειτουργείτε μέσα σε ένα νομοθετικό πλαίσιο ε, για να αντιμετωπίσετε την κρίση. Πρέπει να πάρετε προληπτικά μέτρα και όχι απλώς και μόνο να διαχειριστείτε τα όσα λαμβάνουν χώρα. Ε, θα πρέπει όμως να προσέξουμε τη γραφειοκρατία. Δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε οργανισμούς, ε, ε, υπηρεσίες κτλ. που θα δυσκολέψουν τη ζωή μας αργότερα. θα πρέπει να προβλέψουμε τα προβλήματα και μελλοντικές ε, οικονομικές κρίσεις, αλλά και να επιτρέψουμε στις τράπεζες να λειτουργούν με ένα πιο συντονισμένο τρόπο, με ίδιες συνθήκες σε, όλες, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε διαφάνεια για να γίνουν όλα αυτά και αυτό θα πρέπει οι ρυθμιστές να υιοθετήσουν ε, διατάξεις και διαδικασίες στάνταρτα, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ε, δημοσίευση των αποτελεσμάτων. Ήδη από, το, τα stress test του 2010 είδαμε πόσο σημαντικό, σημαντική είναι η δημοσίευση των αποτελεσμάτων. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα. Ευχαριστώ κύριε Κάντσιαν. Περνάμε τώρα στη διαδικασία και έτσι Κέλλη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Οι τράπεζες ήταν σεβαστές κάποτε στην Ιρλανδία, τώρα είναι μισητές. Και δεν χρειάζεται να εξηγήσω γιατί. Εγώ είμαι εδώ για να δώσω ερωτήσεις, για να κάνω ερωτήσεις και όχι να δώσω απαντήσεις. Πρώτον, όλες οι τράπεζες πρέπει να περάσουν αυτό το τεστ. Δεύτερον, μπορούμε να είμαστε σίγουροι πως από εδώ και μπρο θα αντικατοπτρίζει σε αυτό την πραγματική κατάσταση των τραπεζών. Και τρίτον, ποια εξουσία έχει η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή για να επιβάλλει την εξουσία της σε τράπεζες που έχουν υπερεκτεθεί, δρούν ανεύθυνα κτλ. Και τέλος, ο κ. Κοζές αναφέρθηκε στην ανάγκη να μην εξαρτώμεθα από τις υπηρεσίες αξιολόγησης σε εταιρεία αξιολόγηση. Πώς θα γίνει αυτό το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κέλλη, κύριος Σέμκε για ένα λεπτό. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ που μου δώσετε τη δυνατότητα να θέσω ένα ερώτημα και να το πω πολύ γρήγορα. Εάν ε, δεν είχατε εσείς κύριε Επίτροπε ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλάβει δράση, αναμφίβολα σήμερα η κατάσταση στον τραπεζικό τομέα στην Ευρώπη θα ήταν πολύ χειρότερη από ό,τι είναι. Ωστόσο, μεταβάλλεται με δυναμικό τρόπο η κατάσταση. Κάποια προβλήματα σε σχέση με τη ρευστότητα των τραπεζών έχουν ήδη ξεπεραστεί, αλλά ανακύπτουν νέα προβλήματα και εμφανίζονται νέες απειλές. Εξού το ερώτημα που σας θέτω κύριε Επίτροπε πώς θα ορίζατε τους κινδύνους και τις απειλές που συνεχώς ανακύπτουν σήμερα. Πώς θα τις ορίζατε και ποιοι είναι οι κίνδυνοι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο άμεσο μέλλον. Είπα, έχουν ξεπεραστεί κάποια προβλήματα, εμφανίζονται όμως συνέχεια νέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τσέμκε. Κυρία Μαγκίνες έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μην ξεχνάμε πως υπάρχουν άνθρωποι που επηρεάζονται από αυτά τα προβλήματα. Συνάντησα έναν Ιρλανδό προς την ε, Φραγκφούρτη που πήγαινε με ένα εισιτήριο αλέ μόνο στην Αυστραλία, μετανάστευε. Δέχεται η Κομισιόν πως η ζημιά στην αξιοπιστία της Ευρώπης από το πώς τα θαλάσσωσαν στα πέρσινα στρες τεστ οδηγεί τους Ευρωπαίους πολίτες να κοιτούν ανήσυχοι τις ε, τράπεζες και έχει βλάψει την εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ξέρετε οι Ιρλανδικές τράπεζες πέρασαν ήδη το δεύτερο γύρο και η κυβέρνηση έχει κάνει ένα σχέδιο ε, αναδιάρθρωσης των τραπεζών. Μιλάμε για άλλα 24 δισεκατομμύρια που θα απαιτηθούν και καλές επιχειρήσεις πλέον δεν έχουν κεφάλαιο γιατί δεν τους δίνουν οι τράπεζες. Θέλω να ε, το δει αυτό η Κομισιόν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Μαγκίνες. Ε, η κυρία Μπασέσκου τώρα. Ήθελα να σας πω ότι τα προηγούμενα, είπαμε ότι τα προηγούμενα stress test δεν ήταν αποτελεσματικά, δεν ήταν, αποτελεσμα, ε, δεν ήταν επιτυχή. Και αυτό δυσχεραίνει το όλο σύστημα. Ε, θα πρέπει επομένως τα μελλοντικά τέστα να είναι πολύ πιο ε, σαφή και πιο αξιόπιστα όσον αφορά τα αποτελέσματα τα οποία δίνουν. Είδαμε τι έγινε με την Ιρλανδία πέρυσι. Γι' αυτό θα πρέπει ε, και να προσπαθήσουμε να λύσουμε, αν θέλετε, τα όσα προβλήματα παρουσιάζουν τα stress test. Θα πρέπει οι τράπεζες να περνάνε τα, τις δοκιμασίες αυτές. Θα πρέπει όμως και εμείς να εντοπίσουμε ποια είναι τα σημεία ε, τα οποία πρέπει να βελτιώσουμε, πώς θα ενισχύσουμε τα κεφάλαια παραδείγματο χάρη. Ε, πιστεύουμε ότι οι δοκιμές αυτές θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε, όλες, ε, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα τεστ αυτά. Ευχαριστώ για να τελειώσει η διαδικασία και η κυρία Γκάλπελς. Ευχαριστώ. Η σημασία του θέματος αυτού γίνεται σαφής από το ότι υπέβαλαν το ίδιο ερώτημα τρεις βουλευτές στην Κομισιόν η αξιοπιστία της Κομισιόν εδώ πέρα κινδυνεύει εάν δεν αποκαταστήσουμε με τα νέα τεστ ε, την ε, εμπιστοσύνη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή έχουν τώρα μία νέα μέθοδο, αλλά μετά την απάντηση του κυρίου Επιτρόπου εγώ βλέπω κάποια ανοιχτά ζητήματα. Ένα από αυτά είναι παραδείγματο χάρη το εάν θα ληφθούν υπόψη οι διασυνοριακές διοκτησιακές σχέσεις ή τα διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα. Και να μην μείνει εκτός καμία τράπεζα που διακινδυνεύει την ευρωπαϊκή οικονομική λειτουργία. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μπαρνιέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κάθε έναν και την κάθε μία από όσου πήραν το λόγο και τόσο αργά κιόλα. γιατί είναι δύσκολα θέματα και αυτό δείχνει και την ε, επαγρύπνηση και την ευφυΐα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να ερωτήσω την, ε, να, να, σχολιάσω και την ερώτηση της κυρίας Καλπέλσο για τις ευθύνες της Επιτροπής να σας πω ότι τα stress test αυτή τη στιγμή ε, γίνονται μέσα στα πλαίσια και υπό την εποπτεία της νέας αρχής την οποία έχουμε δημιουργήσει βέβαια. Συνεργαζόμαστε με την αρχή αυτή και όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, και αυτή συνεργάστηκε στην προετοιμασία αυτών των, ε, αυτής της νέας σειράς ε, τεστ, όμως η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών είναι η υπεύθυνη. Ε, τέθη μία προφορική γενική ερώτηση για το ποιες είναι οι μελλοντικέ απειλές, οι κίνδυνοι. Καταρχάς μηδενικό κίνδυνος δεν υπάρχει πουθενά, ούτε εδώ ούτε στην οικολογία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλέψουμε το μέλλον. Και ξέρουμε ότι οι αγορές δρούν πολύ πιο γρήγορα από την δημοκρατία, από το χρόνο το δικό μας τουλάχιστον. Ανεξάρτητα από το αν εμείς θέλουμε και προσπαθούμε να προχωρήσουμε γρήγορα. Τώρα, πώς μπορούμε να είμαστε κάπως περισσότερο προστατευμένοι τώρα από ό,τι πριν από τέσσερα χρόνια. Όταν ήρθε αυτή η κρίση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ε, κινδύνευσε να μας παρασύρει όλους. Μέσα στα πλαίσια μιας διακυβέρνησης, μιας διαφάνειας, μιας ευθύνης προσπαθήσαμε να ε, διορθώσουμε ό,τι έλειπε στο παρελθόν μέσα σε αυτό το κύμα του νέου φιλελευθερισμού που κατάκλυσε τον κόσμο από τη δεκαετία του 90. Ε, πολλά καταργήθηκαν με αυτή την ε, ιδέα, την περίεργη ιδέα της αυτορυθμιζόμενης αγοράς. Εμείς σιγά σιγά και υπομονετικά μέσα στα πλαίσια των, ε, της ομάδας των 20 ε, προσπαθούμε να ε, δημιουργήσουμε εκ νέου ένα πλαίσιο, κάποια εργαλεία κυβέρνησης, διακυβέρνησης, ηθικής θα μπορώ να χρησιμοποιήσω τον όρο αυτό, ε, ε, πράγματα δηλαδή τα οποία έλειπαν από το τοπίο των χρηματοπιστωτικών αγορών εδώ και 15 περίπου χρόνια. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ε, τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν η, η απόφαση που πήρατε για να δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών είναι τόσο σημαντική. Γι' αυτό ακριβώς είπα και στον Ζαν Πολ που αναφέρθηκε σε αυτές ε, ε τους οίκους ε, αξιολόγησης ε, ότι εμείς όλα αυτά τα εντάσσουμε στο μεγάλο εργοτάξιο της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης και ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι προσπαθειές μας. Μέσα σε αυτό το ε- εργοτάξιο, μπορώ να χρησιμοποιήσω και τον όρο ομοσπονδία προφανώς. Δεν διστάζω να το χρησιμοποιήσω τον, ε, τον όρο αυτό γιατί πρέπει να ε, χρησιμοποιήσουμε από κοινού να έχουμε μια ομοσπονδία αν θέλετε προσπαθειών. Πρέπει να ξεπεράσουμε ένα, τον απλό συντονισμό. Επίσης ε, υπάρχει και, όπως είπε ο κ. Γκοζές, ε, είναι ανάγκη να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας ε, για τους οίκους αξιολόγησης. Είμαστε στην τρίτη μας προσπάθεια, η μεταρρύθμιση. Και κύριε Γκοζές για το θέμα υπερβολικής εξάρτησης το οποίο θέσατε όσον αφορά την βαθμολόγηση και την αξιολόγηση από τις αρχές Ιουλίου ε, διαγράψαμε πολλές αναφορές ε, όσον αφορά την αξιολόγηση έτσι ώστε να μετριαστεί κάπως αυτή η υπερβολική ε, εξάρτηση των τραπεζών στην αξιολόγηση και όχι των τραπεζών. Είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει. Επίσης αναφέρθηκαν πολλοί βουλευτές τους οποίους και ευχαριστώ που αναφερθήκατε σε όλα αυτά τα θέματα γιατί εκφράζεται μια θέληση να προχωρήσουμε. Επίσης ευχαριστώ που αναφέρετε το τόσο σημαντικό ρόλο στην Επιτροπή Συστημικών Κινδύνων ε, ε, Έπρεπε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις δυσκολίες ε, και για τον συστημικό κίνδυνο σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξάγουμε τα σωστά συμπεράσματα από τα stress test. Βέβαια, το έργο της εξαγωγής συμπερασμάτων αφορά τα κράτη-μέλη περισσότερο, κυρίως αυτά τα εργαλεία, τα backstop, που και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην περίοδο που θα ακολουθήσει τα stress test. Σας είπα ότι όταν δημιουργήθηκαν αυτές οι τρεις αρχές ε, ελέγχου των συστημικών κινδύνων ότι θα δοκιμαστούμε κατά την πορεία. Και αυτό ακριβώς γίνεται. Ο οργανισμός του κυρίου Μπέα κάνει πάρα πολύ, του κυρίου Ένα κάνει πάρα πολύ δουλειά. Οι άλλες... Ε, ο κύριος κύριε ε, Αναφερθήκατε στα τεστ στον τομέα των εταιριών και, η αντίστοιχη, και ο αντίστοιχος οργανισμός προετοιμάζει, ε, όπως το έκανε και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών για τις τράπεζες, προετοιμάζουμε και τεστ και για τις ασφάλισες. Επίσης, ε, για, τα, για το δημόσιο χρέος η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, και δεν πρόκειται να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, είναι αρμόδια να καθορίσει ε, τις δοκιμασίες Δεν μπορώ να πω, να πω σε λεπτομέρειες. Να σας πω όμως ότι είμαστε σε συνεχή διάλογο με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Ο κ. Γκίγκολτ ε, ξέρει ποια είναι τα, τα μαθήματα τα οποία πρέπει να εξάγουμε και από το προηγούμενο κύμα των δοκιμασιών και από αυτό εδώ. Έχουμε όμως τη φιλοδοξία να συνεχίσουμε τον διάλογο, σεβόμενοι βέβαια τις αρμοδιότητες και την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών όπως θέλουμε και οι άλλοι να σέβονται την εξαρτησία της Κομισιόν. Όμως, κύριε Γκίγκολτ, θα πρέπει ε, με ψυχραιμία να εξάγουμε τα συμπεράσματά μας από το, τις δοκιμασίες που θα ολοκληρωθούν τον Ιούνιο και να βελτιώσουμε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών το επόμενο κύμα δοκιμασιών. Ε, κύριε Μάν, αναφερθήκατε στην ρευστότητα, στον κίνδυνο ρευστότητας. Ξέρετε ότι αυτό το δεν αποτελεί τμήμα της δοκιμασίας. Στις αρχές του έτους η Ευρωπαϊκή Αρχή είχε πει ότι θα γίνει μια, ένας θεματικός έλεγχος των κινδύνων στο τραπεζικό τομέα μέσα στα πλαίσια της ε, συστηματικής ε, αξιολόγησης των κινδύνων ε, που γίνεται σε εξαμηνιαία βάση. Ο κύριος Καράς ζήτησε από τους συναδέλφους και από την Κομισιό να εντάξουμε στην, ε, στρατηγική, στην, μελλοντική, στην μακροπρόθεσμη στρατηγική μας και ούτως ή άλλως συμφωνώ απόλυτα και μέσα σε αυτό το πνεύμα με, τις, ε, με την ομάδα μου εργαζόμαστε έτσι ώστε να σας προτείνουμε την, ε, τις νομοθετικές διατάξεις που θα ρυθμίζουν την, αυτή την διακυβέρνηση διακυβέρνηση που αφορά, παραδείγματος την ευθύνη των μετόχων όπως είπε και στην κυρία Φερέιρα προηγουμένως ε, για, την, ε, για το ψήφισμα της τράπεζας και κάτι άλλο το οποίο έχω κατά νου και που είναι ένας από τους λόγους ε, τα αίτια της κρίσης που είναι τα παράλογα μπόνους και οι αμοιβέ ε, που δίδονται διότι ο καθένα έπαιρνε του κινδύνου, ανέλαμβανε κάποιου κινδύνου, ξέροντα ότι το κίνητο τον θα τον πλήρωνε κάποιος άλλος. Λοιπόν, για τα μπόνους και τις αμοιβέ ε, εξετάζουμε το σύστημα, σύστημα ελέγχου και επίβλεψης των αμοιβών αυτών που είναι ανεπαρκές ούτω ή άλλω. και θα προετοιμάσουμε ένα κείμενο το οποίο θα δούμε πώ θα εφαρμοστεί στα κράτη-μέλη και θεωρούμε ότι αυτή, αυτό αποτελεί μία από τις πηγές της κρίσης. Με αυτό την, την ανάληψη παραλόγων κινδύνων, γιατί θα πρέπει να ε, σε κάποια νυφαλιότητα και σε κάποια ψυχραιμία, αν θέλετε, από πλευρά των τραπεζικών. Ο κύριος Φερέιρα, όπως και ο κύριος Λάμπερτς, αναφέρθηκαν στην έλλειψη συνοχής των stress test. Ε, Είπα, σας είπα ότι ήταν ανεπαρκή τα προηγούμενα, οι προηγούμενες δοκιμασίες. Χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη στην εφαρμογή των τεστ αυτών. Γι' αυτό ακριβώς με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και η peer review θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Μέσα στα πλαίσια, μέσα σε έναν αρμονισμένο μάλλον πλαίσιο, ε, είναι κάτι πάνω στο οποίο εργαζόμαστε, έτσι ώστε να έχουμε το για την επίλυση των προβλημάτων γιατί νομίζω ότι ε, θα μπορέσουμε να υποβάλουμε την πρότασή μας πριν από το τέλος του καλοκαιριού. Πολλοί, ο κύριος Γκίψον, ο κύριος Φόρντ, ο κύριος Κατσίν, η κυρία Μπαζέσκου, αναφέρθηκαν σε αυστηρά, αξιόπιστα και διάφανα τεστ μέσα στα πλαίσια αυτής της ε, οικονομικής διακυβέρνησης την οποία προσπαθούμε να οικοδομήσουμε από κοινού, τα τεστ για το 2011 θα είναι πιο αυστηρά, πιο διάφανα, πιο αξιόπιστα από ότι το προηγούμενο κύμα και θα στηριχθούμε ε, στα διδάγματα αυτά τόν τον των τεστ του 2011 έτσι ώστε την επόμενη χρονιά να έχουμε πιο αυστηρά, πιο αξιόπιστα και πιο ε, διάφανα τεστ στον τραπεζικό τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Καθυστερήσαμε λίγο κύριε Επίτροπε. Είναι πολύ